στην πρώτη ανάγνωση και συμπεριλαμβάνεται από το Συμβούλιο ε, στη θέση του. Οπότε θα μπορούν οι συνάδελφοι με καθαρή συνείδηση να ψηφίσουν τις άλλες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λούλινγκ. Έληξε εδώ η τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο. Και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της κυρίας Σίλβια Αντριάνα Τιτσάου ως συντάκτης. Ενεργειακή απόδοση των κτηρίων είναι το θέμα. Ξεκινούμε τη συζήτηση με την εισηγήτρια. Έχετε το λόγο κυρία Τιτσάου για τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, Επιτροπή το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε για μείωση κατά 20% την κατανάλωση ενέργεια ω το 2020 και για μείωση 20% τη ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ στη συνολική κατανάλωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στι 25-26 Μαρτίου 2010 αποφάσισε να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση κατά 20% ω το 2020. Ο οικονομικός τομέα είναι μια από, αναλογή στο 40% της κατανάλωσης ε, και το 26% στην, ε, ε, και στο 32% του συνόλου των εκπομπών. συνεπώς είναι σημαντική η δράση σε αυτό το τομέα. Το, στα ενεργειακώ αποδοτικά κτίρια επιτυχάνεται κατά μέσο όρο 30% περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης χρησιμοποιείται λιγότερο νερό και έχουν μικρότερο κόστος συντήρησης. Θα μπορούσαμε με, τα, ε, με αποδοτικά κτίρια να, ε, μέχρι το 2030 να δημιουργήσουμε 2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή πρότεινε την αδιατύπωση οδηγίας υπέβαλε στις 13 Νοεμβρίου 2008 τη σχετική νομοθετική πρόταση. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση ε, υιοθέτησε τη θέση του. Στις 22 Απριλίου 2009 Κατά τη διάρκεια τη Σουηδική ε, Προεδρία, ε, συνεχίστηκαν οι με το Κοινοβούλιο και τον Νοέμβριο του 2009 καταλήξαμε σε πολιτική συμφωνία για τι τεχνικέ ε, πτυχέ τη νομοθετική πρόταση. Οι βασικέ κύριε αλλαγέ είναι ένα καινούριο άρθρο και, πολλές, και πολλά εκτιμώντα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση. Η Κομισιόν θα εντοπίσει τα χρηματοδοτικά όργανα ε, και μέσα που υπάρχουν και θα υποβάλει προτάσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2011 για τη χρηματοδότηση. Υποβάλει και σχετική δήλωση. Μέχρι το, 2000, μέχρι το 2020 όλα τα ε, κτίρια θα πρέπει να έχουν ε, περίπου μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο και αυτό το όριο, ε, χρονικό όριο είναι δύο χρόνια πριν για τα δημόσια κτίρια. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένοι στόχοι και δράσεις. Η ενεργειακή απόδοση των ε, κτίριων θα εξασφαλιστεί με, ε, με ανακαίνιση των κτίριων και των δομικών του στοιχείων, τα οποία επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση νέες ε, διατάξεις για τα πιστοποιητικά, ε, δυνατότητα ε, έκδοσης επιστοποιητικών για την ενεργειακή απόδοση μεταξύ αυτών και του δίκτυ. Includerea indicatorului de performanță στο πιστοποιητικό του κτηρίου θα μπορεί να αναφέρεται η ενεργειακή του απόδοση ε, που θα, κάτι που θα χρησιμεύει στην πόλη του κτηρίου καθ' ολοκληρώνει κατά τμήματα. Ε, προβλέπεται διαβούλευση με τοπικές, ε, περιφερειακές και εθνικές αρχές. Έχουμε καινούριες διατάξεις για τους ε, ε, ειδικού εμπειρογνώμονες και τους ε, ντόπιου αρχιτέκτονες έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσει και να προβαίνουν σε μελέτες με αυτοματοποιημένα συστήματα προκειμένου να, μειωθεί, να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση. τα κράτη-μέλη πρέπει να καταρτήσουν στο Ιούνιο 2011 εθνικά σχέδια δράσης για να τηρηθούν οι απαιτήσει ε, που τις οδηγίες για τη μείωση των ε, νομικών φραγμών και φραγμών της αγοράς και την ανάπτυξη νέων οικονομικών και φορολογικών μέτρων. Όλα αυτά βασίζονται στη Συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου από το 2009. Σας συστήνω να το υιοθετήσουμε. Ο Επίτροπος ο κύριος ε, Oettinger. Herr Präsident, Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σπάνια στην ε, πολιτική είναι οι λύσει win-win. Μία τέτοια περίπτωση έχουμε σήμερα μπροστά μας. Η έγκριση της ε, νέας ε, οδηγίας για ενεργειακή απόδοση των κτηρίων για τα κτίρια. Για 40% της, εκατό της ενέργειας κατανάλωσης ενέργειας ε, και για ένα 32% του συνόλου των εκπομπών ευθύνονται τα κτίρια. Οπότε μπορούμε να επιτύχουμε έτσι τους στόχους του 2020 ε, για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και τη μείωση κατανάλωση ενέργειας. Ταυτόχρονα ενισχύουμε την ενεργειακή μας ασφάλεια και δημιουργούμε ανάπτυξη και θέση εργασία στον τομέα των οικοδομών. Επίσης η νέα αυτή οδηγία συνεισφέρει στο ότι οι εθνικοί οικοδομικοί κανονισμοί θα γίνουν πιο απαιτητικοί και θα βοηθήσουν στη μείωση του κόστους των λογαριασμών των καταναλωτών. Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα είναι η καλύτερη και πιο φτηνή ευκαιρία κατά πολέμησης κλιματικής αλλαγής. Θα αναφέρω τρία στοιχεία της νέας οδηγίας που κατά την άποψή μας αποτελούν μεγάλη επιτυχία. Πρώτα απ' όλα Έχουμε τις εθνικές διατάξεις για ανακαινήσεις και νέα κτίρια, που σημαίνει αυτό εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό ισχύει και για μικρότερα κτίρια κάτω των 100.000 τετραγωνικών μέτρων ωφέλιμου χώρου. Ε, όπως επίσης καλύπτουν εδώ πέρα και ανακαινήσεις, όπως παραδείγματος χάρη αλλαγές ε, παραθύρων. Δεύτερον, αυτό είναι σημαντικό και για τους πολίτες μας και για την πληροφόρηση ιδιοκτητών και ενοικιαστών καθώς θα πληροφορηθούν την κατανάλωση και τη δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας του κτηρίου. Αυτό σημαίνει πως θα φτάσουμε στα κτίρια ελάχιστης χρήσης ε, ενέργειας. Και τρίτον, όλες οι νέες κατασκευές από το 2020 θα πρέπει να πληρούν τον αυστηρότατο κανονισμό σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό σημαίνει πως θα έχουμε εθνικά σχέδια δράσης έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι αυτή η οδηγία, είναι μια επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής. Ευχαριστώ τους βουλευτές την κυρία Τικάου για την καλή συνεργασία τους τελευταίους μήνες και για την εξαιρετικά γρήγορη υιοθέτηση της οδηγίας. Τονίσατε πως είναι αυτή η διατύπωση θα συνεισφέρει μόνο εάν εφαρμοστεί γρήγορα και αποτελεσματικά και υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε στην καλύτερη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων π.χ. το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπου θα μπορέσουμε να πούμε πως ένα 4% του προπολογισμού θα πηγαίνει στην εξοικονόμηση ενέργειας εάν δεν χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη επιπλέον θέλουμε να δούμε τη στήριξη των κρατών μελών στην ανακαίνιση υπαρχόντων κτηρίων καθώς βλέπουμε πως ε, τουλάχιστον 51 ε, εκατομμύρια ευρώ από το Πενθυνικό Ταμείο θα κατευθυνθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαι σίγουρος πως με τη στήριξη του Κοινοβουλίου σήμερα θα επιτύχουμε ένα σημαντικό βήμα και σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κύριε πίτροπε. Εξ των πολιτικών ομάδων τώρα οι ομιλητές. Ο πρώτος είναι ο κύριος Ρούμπικ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Τικάου, σας συγχαίρω για αυτή την έκθεση. Είναι ένα μεγάλο βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Έχουμε πάνω από 160 εκατομμύρια κτίρια στην Ευρώπη και τα κτίρια αυτά πρέπει να υποστούν μια θερμική ανακαίνιση για να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια και να μειωθεί η συνολική κατανάλωση ενέργειας. 40% της ενέργειας πηγαίνει στην θέρμανση των κτήριων. Ελπίζουμε πως ε, ένα 5% της συνολικής ε, κατανάλωσης ε, ενέργειας θα έχει εξαφανιστεί μέχρι το 2020 με αυτές τις ανακαινήσεις, αλλά θα δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας. Χρειάζονται εδώ πέρα να δούμε πώς θα εκπαιδευτούν και οι εργαζόμενοι που και θα οικοδομήσουν τα νέα κτίρια και θα ανακαινήσουν τα παλιά. Χρειαζόμαστε λοιπόν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα εξειδικευτούν σε αυτό τον τομέα γιατί έτσι θα κερδίσουν και οι ίδιοι και θα έχουν υψηλότερου μισθού. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπο να βγούμε από την κρίση, γιατί βεβαίω έτσι έχουμε και νέα φορολογικά έσοδα και βεβαίως ε, θα έχουμε και μικρότερη χρήση ορυκτών καυσίμων και θα χρησιμοποιήσουμε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Θεωρώ πως η υποκατάσταση λοιπόν ε, η υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας θα οδηγήσει σε απτές οικονομίες οπότε αξίζουν τον κόπο αυτές οι επενδύσεις δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε ό,τι κάναμε τις τελευταίες δεκαετίες θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε ξανά να επενδύουμε έτσι ώστε ακριβώς σε καιρούς κρίσης να βγούμε με όσο το δυνατόν λιγότερη γραφειοκρατία επίσης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλτσίτης για 1,5 λεπτό. Καταρχήν, θέλω να συγχαρώ την κυρία Τικάου για τη δουλειά της. Η συμφωνία με, τον, με το Συμβούλιο αποτελεί ποιοτικό άλμα στον τομέα αυτό. Το σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν έγκαιρα το νομοθετικό αυτό κείμενο. Το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην εσωτερική αγορά και στην, στον τομέα της ενέργειας. Η οικοδομή είναι ο τομέας που πιο πολύ εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να κάνει. Και αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα για τις νέες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εκεί υφίσταται ένας πολύ μεγάλος αριθμός παλαιών κτηρίων κάτοικοι αυτών των κτηρίων συνήθω έχουν χαμηλά εισοδήματα και είναι αυτοί που πληρώνουν του μεγαλύτερου λογαριασμού βέβαια. Η εξασφάλιση κτηρίων με σχεδόν μηδενικό ενεργειακό ισοζύγιο ε, σημαίνει ε, καινούριε απαιτήσει από τι ε, οικοδομικέ εταιρείε. Είναι ένα φιλόδοξο στόχο. Ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθεί στην πράξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Χολ για τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα θα συγχαρώ την κυρία Τσικά που πραγματικά εργάστηκε άοκ να αφοσιώθηκε στο θέμα. Καθυστερήσαμε πολύ λόγω των αναγκαίων νομικών προσαρμογών που απορρέουν τη τη Αβώνα και αυτό σημαίνει ότι εξεπέμφθη πολύ περισσότερο δεξιού του άνθρακο από ό,τι εξεπέμπεται αν μπορούσαμε να κινηθούμε ταχύτερα μακρά η περίοδος κοίησης του θέματος και φαίνεται να λησμονούμε ότι κάποια από τα στοιχεία που περιέχονται ε, θεωρούνται πολύ ριζοσπαστικά όταν είχαν τεθεί στην αρχή. Κυρίως η κατάργηση του κατοφλίου των χιλίων μέτρων που είχε ε, αναφερθεί στην αρχική πρόταση του Συμβουλίου για το σχέδιο, το σχέδιο του για την ενεργειακή απόδοση. Και ε, μετά σχεδόν να έχουμε κτίρια με σχεδόν ε, μηδέν ενεργειακή απώλεια μέχρι το 2021. Δυστυχώς αυτή η νέα απέτηση για τα νέα κτίρια δεν θα μας βοηθήσει όσον αφορά τους στόχους του 2020. 2020 διοτι όλο και περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο μείωση τουλάχιστον 30% των αερίων του θερμοκηπίου. Και για να έχουμε αποτέλεσμα όσον αφορά τους στόχους στην αλλαγή του κλίματος, τα υπάρχοντα κτίρια είναι αυτά που θα πρέπει να αποτελέσουν στόχο και τις απαιτήσει που θα πρέπει να επιβάλλουμε όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε αυτά. Τρεις βασικές δράσεις θα πρέπει να εξετάσουμε, μάλλον να εφαρμόσουμε αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στα υπάρχοντα κτίρια. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει μια μεθοδολογία πολύ στερεά για την καινοτομία και τη βελτιστοποίηση του κόστους. Πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια, αλλά βλέπετε είναι απαραίτητο αυτό γιατί ήδη έχουμε σπαταλήσει πολύ χρόνο και θα είναι το 2014 μέσως, μέχρι ότου εφαρμοστεί αυτή η μεθοδολογία που θα βασίζεται στην βελτιστοποίηση του κόστους. Θα πρέπει να υπάρχουν αιτήσει εθνικοί στόχοι για την βελτίωση απόδοση των κτηρίων τους κατά συγκεκριμένο ποσοστό. Αν είχαμε δεσμευτικό στόχο ευρωπαϊκό για την ενεργειακή απόδοση, είμαι σίγουρη ότι τελικά θα αναλαμβανόταν αυτή η δράση τάχιστα στα κράτη-μέλη, διότι θα καταλάβαινε τα κράτη-μέλη ότι ένας από του ευκολότερου τρόπου για να πετύχεις ένα στόχο ενεργειακής απόδοσης είναι μέσω συστηματικής αναβάθμισης των υπαρχόντων κτίριων. Και τρίτον, κάτι που είναι ζωτική σημασία στα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν εκ των προτέρων χρηματοδότηση για τη βελτίωση των κτηρίων. Και παρά το έργο του εισηγητού και τις προσπάθειες των σκιωδών, δεν προχωρήσαμε αρκετά όσον αφορά την αναδιάσταση του κειμένου όσο θα θέλαμε από την πλευρά του Κοινοβουλίου και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα να βρούμε χρήματα για την ενεργειακή απόδοση και να μπουν στα προγράμματα οικονομική ανάκαμψη και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην καθυστερήσει όσον αφορά τη σχετική τη πρόταση. Και τέλο, θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των στοιχείων που αναφέρονται στο έγγραφο για την όλη εξέλιξη, για το πόσο δεν εφαρμόστηκε κατά το παρελθόν η νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση. Μπορεί τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας διαβεβαιώσει εφαρμοστεί πλήρως και εγκαίρω αυτή η, οδηγία. Ευχαριστώ. για λεπτά. Ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Συγχαίρω την κυρία Τικάου και τους κοιόδης εισηγητές. Χωρίς ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ήταν τόσο επιτυχής αυτή η οδηγία. Στα δυόμιση λεπτά που έχω θα επικεντρωθώ λιγότερο στην οδηγία αλλά στο τι πρέπει να κάνουμε πέρα για να διορθώσουμε τα ασθενή στοιχεία αυτής της οδηγίας δηλαδή τα υπάρχοντα κτίρια. Τι θα γίνει. Αυτό το οποίο θα χρειαζόμασταν από την Κομισιόν είναι μια πρωτοβουλία που θα κάλυπτε, θα είχε τέσσερα σημεία. Πρώτα απ' όλα βοήθεια στις εθνικές κυβερνήσεις για την εφαρμογή. τελευταία οδηγία δεν εφαρμόστηκε σωστά. Εσείς κύριε Έτιγκερ στη γενική σας διεύθυνση έχετε έναν ολόκληρο υπαλλήλο ο φεύγει τον Ιούλιο. Τι θα κάνετε από πλευράς προσωπικού για την εφαρμογή. Δεύτερον, αναφέρθηκε μοντέλα χρηματοδότησης, τι μπορούμε να κάνουμε στην Κομισιόν για να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα κονδύλια του Περιφερειακού Ταμείου και το τι θα απομείνει επίσης από τα προγράμματα αναζωογόνηση οικονομίας. Τρίτον, χρειάζεται μεγαλύτερη αποδοτικότητα της εργασίας στην οικοδομή. Οπότε χρειάζεται κατάρτιση. Πιο εξειδικευμένοι εργάτες θα αυξήσουν την παραγωγικότητα, αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει πως και οι μισθοί που υπάρχουν σήμερα στην οικοδομή στην Ευρώπη θα αλλάξουν. Οπότε θα πρέπει η Κομισιόν να αναλάβει μια πρωτοβουλία κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ συνδικάτων και εργολάβων και χρειαζόμαστε στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης να δώσουμε περισσότερο βάρος στα κτίρια, τα νέα κτίρια να είναι πιο φτηνά από πλευράς ενέργειας και το σημαντικότερο νέες μορφές οργάνωσης της ανακαίνησης γιατί μπορούμε να χτίσουμε και να ανακαινήσουμε φτηνότερα εάν όλη η ανακαίνιση γίνει καλύτερα και διαμορφωθεί καλύτερα και αυτό πρέπει να ε, ενισχυθεί νομίζω με ευρωπαϊκά ερευνητικά κονδύλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Φόρντ για δύο λεπτά. Και εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Τικάου και τους άλλους εισηγητές για τον τρόπο με τον οποίο έτυχε διαπραγμάτευση σε αυτή η οδηγία. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό μας το θέμα και είναι ευχάριστο που ξεκίνησε η συζήτηση και στα επόμενα βήματα πλέον. ορίζω αυτή την έκθεση. 40% της ενέργειας μας καταναλώνεται στα κτίρια. Συνεπώς χρειαζόμαστε πιο βιώσιμη διαμονή, όχι μόνο εξαιτία των περιβαλλοντικών προβλημάτων του άνθρακα, αλλά και εξαιτία ε, των αυξημένων τιμών της ενέργειας και της, ε, το, του προβλήματο της ασφάλειας της τροφοδοσίας. Είναι, υπάρχουν εθνικές διατάξεις, ε, ήδη σε ορισμένα κράτη και ελπίζω ότι αυτή η οδηγία θα οθήσει και τις υπόλοιπες χώρες να υιοθετήσουν τέτοιες διατάξεις. Είναι σημαντικό να κάνουμε οικονόμηση εκεί που μπορούμε να κάνουμε ε, με καινούρια κτίρια ή με ανακαινήσεις παλαιότερων κτηρίων. Επίσης, οι ιδιοκτήτες και οι εργολάβοι θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Η αναδιατύπωση αυτή έγινε γιατί η αρχική οδηγία δεν είχε η υλοποιηθεί σωστά, δεν έχει εφαρμοστεί σωστά. Συνεπώ θα πρέπει να προσέχουμε πώ θα, εφαρμόσουν και αυτήν την οδηγία τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν θα πρέπει παρακαλώ να βοηθήσει έτσι ώστε οι καλύτερες πρακτικές να γίνουν πιο γνωστές ε, στα κράτη-μέλη και να εξασφαλιστεί ότι τα οι ελάχιστες προδιαγραφές ενεργειακής ε, απόδοσης θα είναι συμβατέ μεταξύ τους. Είναι μεγάλη πρόκληση η εξοικονόμηση ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό ε, και ο δημόσιο και ο ιδιωτικό τομέα να αναγνωρίσει και να δει τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από, τις, ε, από την εξοικονόμηση ενέργειας. Περιβαλλοντικά και οικονομικά ωφέλη. Μια προειδοποίηση όμως. Έχω ένα παράδειγμα στη δική μου χώρα. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, ε, φοβόμαστε μήπως ε, προσθέτουμε πάρα πολύ γραφειοκρατία χωρίς να εξασφαλίζουμε μεγάλη, ε, μεγάλο όφελος από αυτό το μέτρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια κρίση ταυτότητα. Συνεπώ, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχουν θέματα, τουλάχιστον όπω αυτό, στο, στα οποία έχει εξασφαλιστεί συνένεση και κοινή βούληση και αποφασιστικότητα. Αυτό ισχύει από παλιά άλλωστε για αυτό το θέμα. Ας δώσουμε το μήνυμα ότι είμαστε ισχυρότεροι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, όταν συσπηρωνόμαστε γύρω από ένα κοινό συμφέρον. Η κυρία Ματίας για ένα λεπτό. Και εγώ θα ξεκινήσω συγχαίροντας την εργασία και την επιμονή της κυρίας Τικάου. Ήταν ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εργασία της για μια Ευρώπη πιο βιώσιμη. Η ενδιακή δαπάνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ υψηλότερη από το αποδεκτό επίπεδο. Σημαντική λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία. Ήρθε η στιγμή να ακολουθήσουμε μια φιλόδοξη πολιτική και αυτή την πολιτική να τη συνοδεύσουμε με συμπληρωματικά μέτρα. Ιδιαίτερα δεδομένη τη περίοδου κρίσεως που ζούμε. Η οικοδομή είναι ένας από τους ε, κλάδους όπου μπορούμε να δούμε τη ε, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Εκεί μπορούμε να εφαρμόσουμε κρατικές ε, πολιτικές εξοικονόμηση ενέργειας και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να υποφεληθούμε της ευκαιρίας για να επενδύσουμε στη στην βελτίωση της ενεργικής απόδοσης των κτηρίων γιατί είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει και εκατομμύρια θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια. Δεν μιλώ μόνο για τα καινούργια κτίρια, αλλά και για την ανακαίνιση παλαιότερων κτίριων. Ας επωφεληθούμε λοιπόν αυτή τη οδηγία για να αναθερμάνουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Ας γίνουν επενδύσεις οι οποίες είναι στρατηγικής φύσεως και θα μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε και την κρίση. Ελπίζω τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν να επωφεληθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκα για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ξεκινώντας θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση εντόπισε το πεδίο εφαρμογής για την εξοικονόμηση ενεργείας στα κτίρια μέσω βελτιώσεως της μόνωσης και και μόνωση των εξωτερικών τείχων των κτίριων. Εκεί μπορούμε να πετύχουμε μεγάλες οικονομίες. Όμως, δεν είναι μόνο θέμα θέρμανσης, είναι επίσης και το θέμα της θέρμανσης του νερού και το θέμα του κλιματισμού. Νομίζω ότι η οικονομία σε αυτό το τομέα θα είναι πιο δύσκολος. Έχουμε, μάλλον χρειαζόμαστε αρκετά προθυμένα συστήματα, περίπλοκα συστήματα, τα οποία θα πρέπει να μπορούν να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία σε διάφορα τμήματα ενός ε, συγκεκριμένου κτηρίου. Κάθε κτίριο θα πρέπει ε, να εξετάζεται ε, ξεχωριστά και αυτό ισχύει και για τις επιχειρήσεις και για κατοικίες. Ένα κομμάτι λοιπόν, ένα τμήμα των στόχων μας θα πρέπει να είναι και αυτό. Η βελτίωση των προδιαγραφών όσον αφορά τα κτίρια, το σχεδιασμό των κτιρίων, πρόθεση των ευφυών λύσεων για τα διάφορα κτίρια. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα ούτω ώστε οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό των οικοδομών των κατασκευών να βελτιώσουν τι ικανότητέ του και τι δεξιότητε. Ελπίζω να λειτουργήσει, αλλά νομίζω ότι σε πολλού τομεί θα έχουμε δυσκολίε. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρβάλο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ο τομέας των οικοδομών της οικοδομής καταναλώνει το 40% της ενέργειας και εκπέμπει το 30% του συνόλου των εκπομπών. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα έτσι ώστε το 2020 τα νέα κτίρια να έχουν μηδενική κατανάλωση εάν είναι δυνατόν, ή να είναι κοντά στο μηδέν και θα πρέπει και τα παλαιότερα κτίρια να ανακαινιστούν έτσι ώστε να καταστούν ενεργειακά η φόρα. Αυτό θα μειώσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ελπίζω ότι θα δημιουργήσει και νέες θέσεις απασχόλησης. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει γρήγορη βελτίωση του οικολογικού χαρακτήρα των κτηρίων, κάτι το οποίο όπως είπα θα τονώσει και την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται και ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Θέλουμε οι ιδιωτικές και οι δημόσιες επενδύσεις να προχωρήσουν από κοινού και να βοηθήσουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θέλουμε επίσης ε, προγράμματα κνέου ε, κατάρτισης ε, των τεχνητών και των ειδικών που ασχολούνται με το συγκεκριμένο τομέα. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει σωστά τα περιφερειακά ταμεία. Και θα χρησιμοποιήσει τα ταμεία αυτά ως καταλήτες έτσι ώστε να προσελκυστεί ε, ένα νέο κύμα θα έλεγα ιδιωτικών επενδύσεων και να βελτιωθεί η οικολογική αποτελεσματικότητα. ως Παντάρ, ένα λεπτό. Κυρίες και κύριοι, η έκθεση της κυρίας Τσικάου είναι από τη σημαντικότητα τα σημαντικότερα εργαλεία πολιτική στον τομέα του κλίματο και τη ενέργεια που θετήσαν τελευταία χρόνια. Συγχαίρω όλου που συμμετείχαν στη σύνταξη τη εκθέσεω, όλο ιδιαίτερα βεβαίω την εισηγήτρια, την κυρία Τσικάου. Δεν θα επαναλάβω τα ήδη υποθέντα, θα αναφέρω δύο πράγματα. Καταρχά, η οδηγία προσφέρει νέε επιχειρηματικέ ευκαιρίε για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων θα υπάρξει ανάγκη για νέες τεχνολογίες θα υπάρξει και μεγαλύτερη ζήτηση στο μέλλον για υλικά, για οικοδομές που θα είναι πιο φιλικά προ το περιβάλλον, να μειωθεί η χρήση των πόρων, να είναι ανακυκλώσιμα τα υλικά, να κατασκευάζονται ευφυή κτίρια. Οι επιχειρήσεις λοιπόν της Ευρώπης θα ωφεληθούν. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη να επενδύσουν σε τεχνολογίες που μειώνουν της, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των κτηρίων. Τα κτίρια χρησιμοποιούν 40% της ενέργειας Ευρωπαϊκής Ενώσεως και παράγουν 38% των κομμών διοξιδίου του άνθρακος. Και, και χρειάζονται πολλούς πόρους. Δεν ξέρω ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά όμως. Παραδείγματος χάρη η οδηγία περιέχει πρόταση σύμφωνα με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει χρήματα από τα θετικά ταμεία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Εγώ πιστεύω ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να εξευρεθεί από τις υφιστάμενες δημοσιονομικές πολιτικές. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντέλη για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι θετική αυτή η οδηγία. Τη χαιρετίζω, διότι είναι κατεπίγον να καταπολεμήσουμε την αλλαγή του κλίματος. Το 2010 είναι η χρονιά τη καταπολέμησης φτωχίας και του κοινωνικού αποκλεισμού 100, ανάμεσα 50 και 125 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που από μια ενεργειακή ανασφάλεια. Σύμφωνα όμως με τη η νέα νομοθεσία αφορά μόνο τα νέα κτηρία και αφορά τα 2,7 εκατομμύρια νέε κατοικίε το χρόνο, ενώ έχουμε 200 εκατομμύρια παλιές κατοικίε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, θα πρέπει τουλάχιστον να ανακαινιστούν τουλάχιστον 500 εκατομμύρια κτίρια μέχρι το 2050 για να πετύχουν το στόχο. Κύριε Επίτροπε, από το 2007 4% των πόρων ΦΕΝΤΕΡ είναι επιλέξιμα για τη βελτίωση ενεργικής απόδοση των κτιρίων. Αλλά είναι μόνο εν μέρη χρησιμοποιηθέντα αυτά τα χρήματα. Πώς μπορείτε να πιέσετε τα κράτη-μέλη για να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι, διότι διαφορετικά θα εξαφανιστούμε το 2013, ενώ κάποια, κανονικά κάποια ποσά θα πρέπει να αυξηθούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιόμπρο είναι εδώ, λέει ο πρόεδρος, όχι, ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Σάντοργας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος, κύριε Σάντουργας. Κύριε Επίτροπε, όπως προείπαν διάφοροι συναδελφοί, αναζητούμε τώρα τον πιο οικονομικό τρόπο, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε αυτή την καινούργια οδηγία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φρεσκάρουμε το ισχύον νομοθετικό καθεστώς και ευχαριστώ τον εισηγητή, αλλά και τους ε, άλλους συναδέλφους οι οποίοι συνεργάστηκαν. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα κτίρια όπου υπάρχουν πολλές δυνατότητες όχι μόνο για εξοικονόμηση ενέργεια, αλλά και για δημιουργία θέσεων απασχόλησης αλλά επίσης έτσι μπορούμε να εφαρμόσουμε καινούργιες τεχνολογίες. Ξέρετε στην ε, Λιθουανία, τη χώρα μου, πάνω από 80% των εταιριών είναι ηλικία άνω των 20 ετών, οπότε είναι αναποτελεσματικά ενεργητικά. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η οδηγία ήρθε την κατάλληλη ώρα και είναι πάρα πολύ α, πρόσφορος τρόπος να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση και νομίζω ότι στο Συμβούλιο η πρόταση θα συγκεντρώσει την συνένεση, λαμβάνεται υπόψη και η επικουρικότητα μπαίνουν κάποια ελάχιστα πρότυπα για τα καινούργια κτίρια, για τα κτίρια τα οποία έχουν φρεσκαριστεί και έτσι έχουμε όλες τις ε, συνθήκες που αναζητούμε, όλους τους τρόπους που θέλουμε, ώστε να ε, κάνουμε εξοικονόμηση ενεργεία, να εξοικονομήσουμε και χρήματα και βέβαια θα πρέπει ταυτόχρονα να δούμε με ποιες διατάξεις θα ενθαρρύνουμε τον κόσμο να αλλάξει συνήθειες, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, επανειλημμένα αναφέρθηκε, αλλά θα ήθελα να επισύρω και την προσοχή σας εις ότι η επιτυχία της οδηγίας θα εξαρτηθεί εν, εν πολλής εις πόσο γρήγορα θα την αναδεχθούν τα κράτη-μέλη. Οπότε χρειαζόμαστε και αντίστοιχα μέτρα στήριξη. Οικονομικά και από τα κράτη-μέλη και από την Ένωση. Η ενεργειακή αποτελεσματικότητα είναι μια από τι προτεραιότητέ μα. Και γι' αυτό και έχει γίνει και για όλη την Ένωση με προτεραιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch the Eye. Για ένα λεπτό ο καθένας. Πρώτος ο κύριος Μαρινέσκου για ένα λεπτό. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η οδηγία όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα των εταιρείων άμεσα θα έχει επιπτώσεις ή στον κατασκευαστικό τομέα. Θα εξοικονομήσουμε ενέργεια και επίσης θα υπάρχει αντίκτυπος στις ε, αγορές. Θα έχουμε θέσεις απασχόλησης και θα έχουμε περισσότερη ενεργειακή αυτονομία και ασφάλεια της Ένωσης. Πρέπει βέβαια να έχουμε και συνοδευτικά μέτρα οικονομικά, χρηματικά, γιατί αυτός ο εξοικονισμός δεν γίνεται μόνο από τα κρατημέλη. Βέβαια, το μάξιμουμ ποσό το οποίο το Αναπτυξιακό Ταμείο μπορεί να μας δώσει δεν είναι επαρκές, πρέπει να αυξηθεί και θα πρέπει επομένω η Κομισιόν να βοηθήσει και να υπάρξει τελικά αυτό το ταμείο ε, που θέλουμε να συγκροτήσουμε και να σχηματοδοτείται από την ε, ΕΤΕ ε, και από τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται επομένως ένα τέτοιο πρόγραμμα ΕΦΙΕΣ, και να εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη και οι καλές, σωστές πρακτικές να βιωθούν παντού. Να έχουμε τεχνική αρρωγή, αλλά και είπαμε και τα χρηματοοικονομικά μέσα τόσο ώστε να είναι πιο αποτελεσματικά τα κριτήριά μου. για ένα λεπτό. Το. Gratulálok Tikau asszony jelentéséhez és az irányelvhez. Ugyanakkor ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια αλλά η έκθεση αυτή δεν έχει μεγάλη αξία εάν δεν επανδρωθεί με ε, οικονομική υποστήριξη διότι στον ε, προϋπολογισμό μετά από το 2013 και στο Ταμείο Συνοχής πρέπει να κινητοποιηθούν ε, κονδύλια και επιπλέον θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και το ιδιωτικό κεφάλαιο και θα πρέπει να προωθήσουμε διάφορα θέματα κατόπιν αυτού θα έπρεπε να δούμε τι ε, ε, ε, εμπειρίες έχουμε μέχρι στιγμής διότι στην Ουγγαρία έχουμε 250.000 ε, κτίρια τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί και μπορούμε εις, ε, τη, τα κτίρια αυτά να ε, επιτύχουμε πολύ καλή απόδοση αλλά αυτό θα πρέπει να μπορέσει να επεκταθεί και συνήπεδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι καταρχήν η δυνατότητα εξοικονομήσεως ενεργείας στις κατοικίες στο μέλλον είναι αμφισβητήσιμο και η εξυγίανση μπορεί να κοστίσει πάρα πολύ. Άρα δεν έχει καμία αξία ε, να ε, εξυγχρονίσει κανείς κτίρια τα οποία μετά θα παραμείνουν άδεια διότι το ενίκιο θα είναι υπέρογγο. Ε, θα πρέπει λοιπόν ε, παραδείγματο χάρη να ε, υπάρξει μία υποχρέωση για χρησιμοποίηση, δεν θα πρέπει να υπάρξει μάλλον καμία χρησιμοποίηση και επιβολή υποχρεωτικής ηλιακής ενεργείας ή άλλων εξυγχρονιστικών μέτρων διότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ κακή παροχή ε, ενέργειας και ε, ενδέχεται να υπάρξουν επικαλύψεις. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες δημιουργίας ε, εχμών των τιμών διότι δεν έχουμε ακόμη τα αναγκαία μηχανήματα για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα. Ε, χαιρετίζω και εγώ την ε, πρόταση αυτή και πιο συγκεκριμένα κάτι το οποίο είπε πολλοί συνάδελφοι για τα κτίρια που είναι σαφές ότι όπως έχει η κατάσταση θα πρέπει λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση να είμαστε σίγουροι ότι τα κτίρια αυτά θα είναι στη θέση του το 2050 Άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι για, για αυτά τα κτίρια, γιατί ξέρετε υπάρχει κρίση και στη δική μου χώρα και ε, από τη μία μεριά υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη στέγαση, από την άλλη μεριά υπάρχουν χιλιάδες ε, κενών. Επομένως ε, θα πρέπει να φροντίσουμε γιατί θα πρέπει να καλύψουμε την ανάγκη αυτή για περισσότερη στέγαση, να επικεντρωθούμε αντί να χτίσουμε καινούργια στα υπάρχοντα. Και αυτό θέλω να πω κύριε Επίτροπε, ότι θα πρέπει οι κυβερνήσει να χρησιμοποιήσουν το διαρθρωτικό ταμείο για το πρόβλημα αυτό και να γίνει χρήση του ταμείου ευθύ αμέσω γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η υπόθεση. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πριν από οτιδήποτε άλλο να συγχαρώ την, τον εισηγητή γιατί έχει κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δουλειά. Είναι αλήθεια ότι τα κτίρια έχουν ε, πολλές δυνατότητες βελτίωσης και αυτό είναι θα έλεγα και ένας από τους στόχους ε, τους οποίους θα πρέπει να έχουμε στην πολιτική του 2020. Τα πιστοποιητικά ενεργειακής αποδοτικότητας είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να πληροφορείται ο πιθανός αγοραστής. Στη χώρα μου έχουν υπάρξει προσπάθειες να υιοθετηθεί αυτή η μέθοδος της έκδοσης ε, ε, των πιστοποιητικών των ενεργειακών ήδη από φέτος, αλλά υπήρξε μια αναβολή λόγω της έλλειψης εκτιμητών. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το αργότερο στις αρχές Ιανουαρίου του 2011 θα αρχίσει η έκδοση των ενεργειακών πιστοποιητικών. Αυτό θα μειώσει τα κοινόχρηστα, θα μειώσει το κόστος των λογαριασμών κοινή ωφέλεια και είναι γενικότερα κάτι το θετικό και στο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Děkuji, pane předsedo. Není pochyb o tom, že zvýšení energetických úspor budov i díky... Έχουμε αυτή την αύξηση ε, τον, της προσπάθειας για καλύτερη για απόδοση των κτηρίων να είναι το θέμα και πολιτικό είναι θέμα επιθυνότητας γιατί να μπορέσουμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο βιώσιμη και την ανάπτυξη πιο βιώσιμη ούτως ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε το ότι έχουμε μια πολιτική μια πολιτική που πάει προς τα μπρος όσον αφορά την αυτονομία την ενεργειακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε τόσο εξαρτημένοι από φυσικό αέριο αλλά και πετρέλαιο από τις τρίτες χώρες. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη βιωσιμότητα και των νέων ε, κτηρίων και των παλαιών όμως. Βεβαίως ε, πρόκειται για κάποια προσπάθεια που θα χρειαστεί οικονομική υποστήριξη από όλα τα κρατημέλη και έτσι να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Εγώ επομένως επιψηφίζω αυτή την πρόταση και ε, την πρόταση επίσης να έχουμε ένα συγκεκριμένο ταμείο και όχι μόνο για την θέρμανση αυτών των νέων κτηρίων, αλλά να φροντίζει γενικά η ενεργειακή αποδοτικότητα. Βέρτμαν, για ένα λεπτό. Αξιότιμοι συνάδελφοι, το 2008 υποχρεώθηκε και δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει ε, την ε, ε, κατανάλωση ενεργείας στα κτίρια με κτίρια χαμηλής ενεργείας και έτσι δεν θα μειωθεί μόνο η κατανάλωση ενεργείας αλλά θα συμβάλλει και στην επίλυση της κρίσεως και θα δημιουργήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο θέσεις εργασίας εργασίας και ε, θα μπορέσουμε ε, να ενισχύσουμε τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και επιπλέον θα ανακαινιστούν τα, νέα, τα παλαιά κτίρια ε, για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έτιγκερ έχει το λόγο.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 Αξιότιμες ε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, εδώ εξετάζουμε τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων, την ανακαίνιση και την ενεργειακή απόδοση ε, για να μπορέσουμε να μειώσουμε τις ε, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Εάν λάβετε υπόψη και τις πηγές ενεργείας, τους ηλεκτρικούς ηλεκτρικούς σταθμούς και, την, και την αυτοκινητοβιομηχανία βλέπετε ότι υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις ε, ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων στην προσπάθεια αυτή τους οποίους πρέπει να πείσουμε ε, στα κτίρια όμως υπάρχουν αντιμέτωπες πολλές ενότητες πολιτών οι ιδιο ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ή κοινότητες με τα οικοδομικά προγράμματά τους, τα, οι περιφερειακοί παράγοντες οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν τα νέα ε, αυτά συστήματα και ε, όπου πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή επέμβαση και βεβαίως στα κτίρια είναι η πιο σημαντική ε, επέμβαση και υπάρχουν οριζοντίως και καθέτως εκατομμύρια συμμετέχοντες. Γι' αυτό και η οδηγία αυτή είναι ένα πολύ βασικό θέμα σήμερα αλλά δεν είναι η τελευταία και τελική λύση. Γι' αυτό και σημειώνω τις προτάσεις σας, τα σχόλιά σας, τις παρακολούθησα με μεγάλη προσοχή και να είστε βέβαιος ότι για μένα η εφαρμογή της οδηγίας είναι εξίσου σημαντική όσο και η επεξεργασία της διότι η αξία της θα είναι να την εφαρμόσουμε και θα χρειαστεί όλοι οι παράγοντες να συμμετάσχουν τα κράτη, τα κράτη-μέλη, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες των κτηρίων αυτών. Δεν θέλουμε να υπάρξουν μόνο νέα κτίρια αλλά και όταν υπάρχουν ανακαινήσεις να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα μέτρα εξοικονόμησης ενεργείας και γι' αυτό υποβάλλουμε την πρότασή μας για να μπορέσουμε να περιορίσουμε κατά 15 εκατομμύρια ευρώ και ε, την, ε, τις επόμενες εβδομάδες θα υποβάλουμε την τελική μας πρόταση για να δούμε εάν θα υπάρχουν περισσότερες εξοικονομήσεις πέραν των 115 ε, εκατομμυρίων ή λιγότερο ποσό. Μέχρι τον Ιούλιο λοιπόν θα έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή για την αποδοτικότητα των νεοσύμων ε, πηγών ενεργείας και ε, των ε, συμβατικών. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τον συνάδελφο Χάν για να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τα περιφερειακά προγράμματα όσον αφορά τους ενεργειακούς στόχους και θα του τονίσω τις παρατηρήσεις σας επίσης για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο στο πρόγραμμά μας πρέπει να περιληφθούν και τα θέματα των κτηρίων και της ενεργειακής εξοικονόμησης διότι υπάρχει επόμενη περίοδος. Ξέρετε ότι έχουμε μεγάλα προγράμματα στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω τα κράτη-μέλη θα μας αυξήσουν τη χρηματοδότησή τους διότι υπάρχει μία κρίση και άρα θα πρέπει ο προϋπολογισμός μας να περιοριστεί και να μπορέσουμε να ικανοποιηθούμε από αυτή τη συρρήκνωση των μέτρων. Για θα χρειαστεί συγχρόνως να υπάρξει έρευνα για την ανάργεια, προγράμματα για εξοικονόμηση ενεργείας επιτόπου και βελτίωση των υποδομών. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο να συζητήσουμε πώς μπορούμε να εμπλέξουμε τις περιφερειακές τοπικές εθνικές αρχές, οι εθνικές αρχές για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μας ανακαίνησης και να το συμπληρώσουν. Είναι ένα βασικό θέμα και δεν είναι το τελευταίο βήμα. Γι' αυτό και είμαι βέβαιος ότι θα μας ελέγχεται αενάως και θα παρακολουθείτε την εφαρμογή της οδηγίας στην πράξη για να δείτε εάν προχωρά ορθά. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές που παρενέβησαν και πρέπει να σας πω ότι σε άλλες περιοχές του κόσμου ή στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Κίνα παρακολουθούν τις κινήσεις Ευρωπαϊκής Ενώσεως διότι προπορεύεται η Ευρώπη από τις άλλες χώρες και γι' αυτό σας ευχαριστώ doresc să mulțumesc întâi și întâi shadow raportorilor pentru sprijinul Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς και τους σκιώδεις εισηγητής για την υποστήριξή τους. Κύριε Πίτροπε, είπατε κι εσείς ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο οικολογικό των κτηρίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ένας εταίρος σας ο οποίος θα προσπαθήσει να συνεισφέρει με τα του μέτρα και μέσα και κυρίως να προσδώσει διαφάνεια στις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στις λήψεις των αποφάσεων. Οι ευθύνε φυσικά δεν απόκεινται κυρίως στα κράτη-μέλη και νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών η οποία προβλέπεται για το 2010 έτσι ώστε να στρέψουμε περισσότερες ροές, περισσότερες πιστώσεις στην αποτελεσματικότητα την ενεργειακή των κτηρίων. Υπήρξαν κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να μειώσουν και το συντελεστή, θα προβλέψουν και τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τα μέτρα καλύτερης ενεργειακής αποτελεσματικότητας των οικοδομών. Τα μέτρα πρέπει να ληφθούν όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να απορροφήσουμε τα κατάλληλα ποσοστά από πλευράς των περιφερειακών ταμείων, όπως προβλέπονται από το 2010 μέχρι το 2013, και μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσουμε να απαιτήσουμε περισσότερες πιστώσεις για την περίοδο η οποία θα ακολουθήσει το 2013 και η αύξηση αυτή μπορεί να φτάσει το 10%. 815 εκατομμύρια δεν χρησιμοποιήθηκαν πέρυσι και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εφόσον έχουν εξοικονομηθεί στην πρωτοβουλία έξυπνη πόλη, Smart City. Θα πρέπει λοιπόν Αυτές να είναι οι προτεραιότητές μας και φυσικά να δώσουμε και το βάρος που απαιτείται και στην Ήπεθρο, όχι μόνο στις πόλεις μικρές και μεγάλες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τικάου. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαρθεί αύριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση για την έκθεση του κυρίου Μάντερς ονομασίες και συναφείς επισήμανση κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων. Είναι εδώ η εισηγητής. Very good. Ε, τον λόγο έχει ο εισηγητής, ο κύριος Μάντερ